Bene, allora se prendete poco... Εάν επιτρέπετε, καλημέρα σας καταρχάς, να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε να προλάβουν και οι τελευταίοι συνάδελφοι να μπουν, διότι έχουμε καθυστερήσει λίγο σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Η πρώτη πληροφορία που θα ήθελα να σας δώσω είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρα, πρέπει να το ξέρετε όλοι νομίζω, αλλά τέλος πάντων σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση που προβλεπόταν για τις 10 Ιανουαρίου έχει ακυρωθεί. Επομένως 10 Ιανουαρίου δεν θα υπάρξει συνεδρίαση Ήτρε. Ενώ τότε εκείνη την ημερομηνία θα γίνει πρώτος τρίλογος για τον ορίζοντα 2020. Και η επόμενη συνεδρίαση της ΙΤΡΕ θα λάβει χώρα στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που θέλω να σας δώσω. Η δεύτερη πληροφορία είναι ότι χτες οι συντονιστές αποφάσισαν να δώσουν εντολή για την διαπραγμάτευση για το, πρόγραμμα, για, την, για το θέμα Skinner, ε, για την Ευρατόμου και σήμερα έχουμε τρεις ψηφοφορίες. Το, η πρώτη αφορά την έκθεση Μέρκες η δεύτερη την έκθεση Correira de Campos και το, η τρίτη για την, για, το, για την έκθεση Skinner που αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για την εντολή που θα δοθεί. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ας ε, κάνουμε μια δοκιμή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, να δούμε και τις παρουσίες χρησιμοποιήστε το, την κάρτα σας και άρχεται η ψηφοφορία, η δοκιμαστική. Πέρας της ψηφοφορίας έχουμε επαρκή αριθμό παρόντων για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την πρώτη έκθεση. Παλά. Μια Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Μέρκης. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Α, όχι, λάθος. 7. Τροπολογία 7. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ε, συγγνώμη, συμβιβαστική πρόταση 5. Α, πρώτα θα κάνουμε ηλεκτρονική δοκιμή για την τροπολογία, για συμβιβασμό 4. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 21 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Λοιπόν, τροπολογία 32 Grazie. E siccome è stato respinto il compromesso 4, Εφόσον απορρίφθηκε η συμβαστική πρόταση 4, πρέπει να ε, ψηφίσουμε τι επόμενε τροπολογίε, τι οποίε δεν ψηφίσαμε. Επομένω, μετά τη συμβαστική πρόταση 4 που απορρίφθηκε, έχουμε την τροπολογία 9. Υπέρ τη τροπολογία 9, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Λοιπόν, ε, ελέγχουμε την τροπολογία 9. Πέραση ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, το ελέγχουμε. Ε, ψηφίζετε περίπου όσοι υπέρ και τόσοι κατά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την 27 υπέρ. Ε, 21-21. Απορρίπτεται. Τρεοπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, το ξαναελέγξουμε. Τροπολογία 28. Ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Λοιπόν, τη συμβαστική πρόταση 5 την ψηφίσαμε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 με μία προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 και 42 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44, 45, 46 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Πέρες ψηφοφορίας. 20 με 22 απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ελέγχουμε την τροπολογία 24. Πέρα της 21 21-22 απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. 39 υπέρ, 1 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Μέρκης. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση, έκθεση Κορέιρα Ντεκάμπος, υπέρ της, συμβαστικού κειμένου όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορία 37 υπέρ 5 εποχές εγκρίνεται. Ψήφος ε, για, την, ε, για το κείμενο για, ε, νομοθετικού περιεχομένου. Πέρας ψηφοφορίας 38 υπέρ Πέντε αποχές εγκρίνεται. Και τελευταία ψηφοφορία για τις ε, θεσμικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την έκθεση Skinner. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 11 κατά, 7 αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση σχετικά με την πορεία των τριμερών διαλόγων. Se ci sono persone che devono uscire, fatelo nei prossimi due minuti. Αν θέλει κάποιο να αποχωρήσει, το κάνει σε επόμενα δύο λεπτά, παρακαλώ. Το συλλόγο τον έχει συνάδελφο Τσίτσεστερ, ο οποίο θα μα δώσει πληροφορίε ε, σχετικά με την πορεία των τριμερών διαλόγων, σχετικά με την ΕΝΙΖΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για ανεπίσημες ε, διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου για τον ΕΝΙΖΑ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων Πληροφορικής. Έχει υπάρξει μία παύση στις διαπραγματεύσεις λόγω του ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε έναν ικανό αριθμό ετοιμάτων δικών μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συμβιβασμό και αποφασίσαμε επομένω να ξανασυνεδριάσουμε στις αρχές του επόμενου έτους για να κλειδώσουμε τις διαπραγματεύσεις και να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Αν συμφωνείτε λοιπόν, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω αρκεί να πω ότι η πρόοδος έχει επιτευχθεί στις συναντήση που είχαμε με το Συμβούλιο, όχι όμως επαρκής πρόοδος. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αν συνάδελφοι έχουν απορίες, ευχαρίστω να τις απαντήσω. Θα προτιμούσα όμως να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλοι οι σκιώδεις συγητές συμμετείχαν πλήρως σε όλα τα στάδια των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Τσίτσεστερ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Δεν ξέρω, θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι, μήπως έχει κάποια απορία που θα μπορούσε να λύσει ο κύριος Τσίτσεστερ, κάποια απληροφορία. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα ε, θα έπρεπε να ακούσουμε και την ε, ενημέρωση σχετικά με την πορεία των τριμερών διαλόγων για τον Γαλιλαίο, αλλά δεν έχουν το αρμόδιο συνάδελφο. Α, όχι, μισό λεπτό. Εσείς μιλάτε εξ ονόματο πιανού, α, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάρα πολύ ωραία. Α, όχι, δεν σας ήξερα, γι' αυτό ρωτάω, συγγνώμη. Λοιπόν, η Κομισιόν έχει τον λόγο. Εργάζομαι για τη Γενική Διεύθυνση Connect και είμαι υπεύθυνο για την υπηρεσία που παρακολουθεί την υπόθεση ΕΝΙΖΑ. Να επαναλάβουμε την ε, αποφασιστικότητα που θα δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό και υπολογίζουμε και στην ε, καλή διάθεση των ε, συνομοθετών μας και στην διαλλακτικότητά σας για να έχουμε επικοδομητικό τριμερή διάλογο στις αρχές της χρονιάς ώστε να ανανεωθεί και η εντολή εγκαίρως. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι πάνω σε αυτό το θέμα έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Έλμα. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη παρατήρηση, αυτά που ακούστηκαν τώρα μετά όσα είπε ο κύριος Τσίτσεστερ, αλλά εμείς να σας πω ότι υποστηρίζουμε την θέση του ε, εισηγητή ε, στο ΕΛΚ. Δεν είναι θέμα καλής θέλησης, αλλά Ήταν εντυπωσιακό το όλο θέμα του, των τριμερών διαλόγων. Το Συμβούλιο ε, έκανε διάφορες προτάσεις για πολλά αμφιλεγόμενα θέματα. Και δεν ξέρω εάν θυμάται το Συμβούλιο τι ελέγχθη σε αυτόν τον τρίλογο. Επομένως, τα σχόλια της Κομισιό δεν ε, έχουν εμάς αναποδέκτες. Τα σχόλια της, ε, τα σχόλια της Κομισιό πρέπει να τα κάνουν στο Συμβούλιο. Καλώς. Ο, ο συνάδελφος Τσίζες θα να προσθέσει κάτι. Όχι. Επομένως, α, θεωρούμε ότι ολοκληρώνεται η ενημέρωση αυτή. Πιλάρ για τον Γαλιλαίο. Πρόεδρε, η συνάδελφος Μαρία Μαρινέσκου δεν μπορεί να έτσι. Και εκ μέρους της θέλω να πω τα Κατάσταση ως προς την Κυπριακή Προεδρία έχει οδηγήσει στην αποσαφήνιση του κειμένου σε πολλά σημεία. Ε, πρόεδρος, δεν ολοκληρώσαμε Μάλλον, να πω ότι ολοκληρώσαμε την ενημέρωση ότι αφορά το ΕΝΙΖΑ. Εσείς μιλάτε για τον Καλλιλέο; έτσι. Ναι πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τον Γαλιλαίο και τον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Μαρινέσκο με ενημερώνει ότι για την Κυπριακή Προεδρία και τον άτυπο τριμερή διάλογο αποσαφινίστηκε το κείμενο των άρθρων σε πολλά σημεία και για τι αιτιολογικές σκέψει, Μα είπε ότι ο κ. Μαρινέσκου συζητήθηκε ήδη με προσώπους τη Ιρλανδική Προεδρία. συζήτησε τα σημαντικά θέματα για το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι με δύο γύρου των διαλόγων ε, επί Ιρλανδική Προεδρία θα μπορέσει να περατωθεί το θέμα. Αυτή είναι η ενημέρωση που θέλω να σα δώσω. Επί τη αρχής φαίνεται ότι είμαστε εντό ε, προθεσμιών ω προ το χρονοδιάγραμμα και ω προ την πρόοδο που πρέπει να επιτελέσουμε. Ευχαριστώ κυρία Ντελκαστήγιο. Θέλει κανείς το λόγο σε σχέση με την ενημέρωση για αυτά τα δύο ζητήματα. Όχι, ωραία. Έχουμε λίγο χρόνο, 20 λεπτά, για την παρουσίαση της ad hoc ενημέρωσης για την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία δεδομένων και τον αντίκτυπο στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσουν δύο ερευνητές, ο κύριος Κέιβ από την Ραντ και ο κύριος Ρόζενταλ. Um, Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε συντομία την έκθεση για την ε, επίδραση που θα έχει η αναθεώρηση της προστασίας των δεδομένων στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν τη μετατόπιση με τη νέα οδηγία, μάλλον από οδηγία σε κανονισμό. Και μας ζητήθηκε να σας αξιολογήσουμε την επίπτωση που θα έχει αυτό στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Κατά βάση, αυτό μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις, ε, τρία άρθρα μας απασχόλησαν συγκεκριμένα. Το άρθρο 20 για την αυτόματη επεξεργασία και το profiling, το άρθρο 28 για τις ε, αρμοδιότητες του ελεγκτή δεδομένου και το άρθρο 6.1f ε, και 44H1 για την ε, μεταφορά δεδομένων, το data migration. Τις επιχειρήσεις τις βλέπουμε κυρίως ως οικοσυστήματα και βλέπουμε και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εταιριών. Και μετά από τη μελέτη μας καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιες συστάσεις. Θα σας παρουσιάσω. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 20, θα θέλαμε να είναι πιο ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά σε άτομα τα οποία είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μη διαφοροποιημένη προσέγγιση. Στο άρθρο 28 λέμε ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένη η απαιτούμενη τεκμηρίωση και θέλουμε να υπάρχουν για κάποιες ιεραρχίες, ώστε να μπορούν οι ελεγκτές να πιστοποιούν αυτούς που επεξεργάζονται τα δεδομένα και ή μάλλον αντιστρόφως. Ό,τι αφορά το άρθρο 44, δεν νομίζουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ σε σχέση με τα άλλα δύο άρθρα τουλάχιστον. Πρέπει πάντως να είναι για σκοπούς διαχείρισης δεδομένων της υποπαραγράφους α έως ε, γ και για τη συγκατάθεση έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά θέλουμε να είναι η διαχείριση των δεδομένων αποτελεσματική και εκεί νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Βλέπετε ένα heat map που έχουμε φτιάξει εδώ. Έχουμε κάποιες ε, κάποιους τομείς τους οποίους ε, αναλύουμε, τέσσερις συγκεκριμένα και βλέπετε πώς επηρεάζουν τα άρθρα αυτά. Πιο πολύ επηρεάζει το άρθρο 20 όπως βλέπετε. Δεν είναι λοιπόν τελείως ουδέτερη αυτή η πρόταση για τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και μάλλον θα επηρεάσει και τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν. Η σχέση μεταξύ καινοτομίας ανταγωνιστικότητα και ιδιωτικού βίου, ιδιωτικής σφαίρα. Έχετε κάποια πιο αναλυτικά στοιχεία στην αίθουσα. Υπάρχει λοιπόν μια ειδική έκθεση για αυτά τα θέματα, για την σχέση που έχουν οι διατάξεις περί ιδιωτική σφαίρα με την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Τέσσερι μελέτε περιπτώσεων είχαμε κάνει, όπω σα είπα. Σα είπα στο χύπημα από την τέσσερι τομεί που μελετήσαμε. Έχουμε τρει επιλογέ, τρία σενάρια. Η επιλογή 0 είναι ο προτινόμενο κανονισμό, η επιλογή 1 ο κανονισμό με τροποποίηση και έχουμε και μια άλλη επιλογή που θα ήταν ε, η αυτορύθμιση ή συνρύθμιση. Δεν το αξιολογήσαμε όμως στη μελέτη επισήμως. Έχουμε κάποιες βασικές αλλαγές ρυθμιστικές καταρχάς, τις βλέπετε, σε ό,τι αφορά το άρθρο 20. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε και την ε, ορολογία natural person, φυσικό πρόσωπο να λέγεται και όχι data subject. Δεν φαίνεται ποια δικαιώματα έχουν τα φυσικά πρόσωπα και μετά να μιλάμε για δικαιώματα των υποκειμένων των data subjects. Τα group profiles μπορούν να εξαιρούνται, αλλά μπορεί τα individual profiles, τα μεμονωμένα προφίλ να μπουν. Βέβαια θα πρέπει να προστατεύονται και τα συμφέροντα των data subjects. Mr. K. take over. Thank you very much. Επόμενος συνάδελφος τώρα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Άρνολντ. Επειδή, όπως είπατε, δεν έχουμε χρόνο, θα προσπαθήσω να αποφύγω τις πολλές λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τον αντίκτυπο, ε, αλλά θα βρείτε και σχετικά έγγραφα και στο βάθος της αίθουσας με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Και το πρώτο στοιχείο που εξετάσαμε, να πω ότι αφορούσε την διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες με οικονομικά στοιχεία και θα ήθελα εδώ να καταστεί σαφέ ότι η καινοτομία και το απόρριτο επηρεάζονται από τι δυνάμει τη αγορά. Τα επιχειρησιακά μοντέλα που σχετίζονται με την ζήτηση από τους πολίτες για το απόρριτο σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Εάν βρουν τέτοια συστήματα με, απαραίτητη, την αναγκαία προστασία στην αγορά οι πολίτες, το εκφράζουν τα ζητούν και έτσι οι προτιμήσει των καταναλωτών καθαρίζουν και το υψηλό επίπεδο προστασία. Εάν όμω δεν υπάρχει υψηλή προστασία, δεν την αναζητούν κιόλα οι πολίτε, τότε δεν εκφράζεται και αναλόγω η αγορά και δεν χρησιμοποιούνται αυτέ οι υπηρεσίε δεν εξυπηρετούνται ανάγκε των καταναλωτών, αλλά τρίτων μερών που προσπαθούν με, οικονομικό, με οικονομικά βιώσιμο τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτά τα δεδομένα και έτσι πέφτει το επίπεδο τη προστασία. Ζούμε βέβαια σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και οι επιπτώσεις ε, τη προστασία των δεδομένων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπω στις ΗΠΑ που εμπορικέ δυνάμεις επικεντρώνονται πιο πολύ ε, στις ε, δυνάμεις των καταναλωτών, στις ανάγκες των καταναλωτών. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που αξιολογήσαμε είχε να κάνει με την διάσταση της αγοράς. Υπήρχαν τρεις επιλογές με πολύ διαφορετικές επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα το βαθμό στον οποίο οι δυνάμεις της αγοράς καθορίζουν το επίπεδο προστασίας των ευρωπαϊκών εταιριών οι οποίε έχουν πρόσβαση στην αγορά μεν, αλλά μπορούν να προτείνουν και λύσει για όσου ενδιαφέρονται για την εμπιστευτικότητα ανά τον κόσμο. Βέβαια το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχουν και οι ανάλογες αξιολογήσεις. Το δεύτερο θέμα της αξιολογής έχει να κάνει με το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων. Εδώ το όλο θέμα είναι η συνένεση, η συγκατάθεση. Εάν υπάρχει τεκμηριωμένη συγκατάθεση και αν ασκείται μας απασχόλησε, είδαμε ότι η τιμή είναι διαφορετική για ε, ε, τους ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες του κόσμο, όπως στις ΗΠΑ για διάφορες υπηρεσίε ε, αυτό καθορίζεται από τι εταιρείε. Αλλά πολλές φορές η συγκατάθεση, η δυνατότητα συγκατάθεσης ε, δεν ισχύει πλέον ε, χωρί να ενημερώνεται καν ο καταναλωτής. Στην Ευρώπη πολλές φορές τα άτομα, οι πολίτες δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν, δεν ενημερώνονται. Αλλά πολλές φορές ο στόχο ακριβώ θα πρέπει να είναι η προστασία των δεδομένων, καλύπτοντα τι ανάγκε των πολιτών. Εντάξει, έτσι. Option the self-regulation or co-regulatory option, is sort of the least... Η επιλογή 2, το βλέπουμε και το είδαμε προηγουμένως, είναι το θέμα για την, αποδο... για την αποτελεσματικότητα. νομίζει και η ίδια η βιομηχανία ότι μπορεί να κάνει, η ίδια η αγορά. Αλλά Σίγουρα για τον περιορισμό του κόστου πρέπει να υπάρχει και ευθυγράμμιση με, την, ε, με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα τα συμπεράσματά μα. Οι επιπτώσει στην αγορά ξεπερνούν αυτού που περιλαμβάνει η μελέτη αντικτύπου, είναι και οικονομικού χαρακτήρα. Έπειτα υπάρχει μια αποτιθέμενη ε, διάσταση μεταξύ τη εμπιστευτικότητα και τη καινοτομία, αλλά πολλοί υπεύθυνοι τη καινοτομία καταλαβαίνουν τι θα πει εμπιστευτικότητα και υπάρχει και ένας αλληλοσχετισμός. Και έπειτα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη το παγκοσμιοποιημένο σκηνικό, ε, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Διότι υπάρχουν ανταγωνιστικέ δυνάμει στο ευρωπαϊκό τοπίο, αλλά υπάρχει δυνατότητα συνεργασία και από τι δύο πλευρέ. Υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα για τα τρία άρθρα και στου τρει τομεί, αλλά για σκοπού οικονομία του χρόνου δεν θα τα παρουσιάσω τώρα. Εάν θέλετε μπορούμε να τα θίξουμε στις ερωτήσεις σας. Τέλος, σε ό,τι αφορά την προτιμόμενη επιλογή που ε, προκύπτει και από τις συστάσεις μας, η, επιλογή, ε, η πρώτη επιλογή θα έδινε ισχυρά, ισχυρά κίνητρα στους ξένους επενδυτές να, και παροχής υπηρεσιών να παρουσιάσουν ε, τις στρατηγικές τους και στην ευρωπαϊκή αγορά Επίσης δημιουργείται βάση για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ισορροπίας στην ε, προστασία των δεδομένων. Τώρα σε σχέση με το άρθρο 20 υπάρχουν νέες τεχνικές όχι μόνο για την προστασία της εμπιστευτικότητας αλλά και για την εξέβρεση σωστής ισορροπίας ε, προστασίας των δεδομένων. Ο, ο κανονισμός όπως τώρα προτείνεται θα επέτρεπε να επιταχυνθεί η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήταν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση ή να εκφράσει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν ξέρω, θέλει κανείς να πάρει το λόγο για όσα για τις ενημερώσεις που ακούσαμε. Αν όχι, ευχαριστούμε τους δύο εισηγητές. Λοιπόν, δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Η κυρία Νίμπλερ, συστήσατε πάρα πολλά ζητήματα και με τέτοια ταχύτητα που τα είπατε, βέβαια δυσκολευτήκαμε να συγκρατήσουμε και πολλά. Προτείνεται νέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και ο πρώτος ομιλητής μας είπε για τρία άρθρα, το 20, το 28, το 44, παράγραφο ένα συγκεκριμένα και πώς αυτά επηρεάζουν. Και για τις επιπτώσεις μας είπατε εσείς και είπε και ο συνάδελφός σας κάποια άλλα πράγματα. Και οπότε καταλάβαμε με τον κανονισμό αυτό, αν τεθεί σε ισχύ, θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις. Και για τη βιομηχανία, για τον κλάδο αυτό στην Ευρώπη. Αλλά συγκεκριμένα τι λέτε. Πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό τη μοντέλο εντελώ οι μικρέ επιχειρήσει. Και από τεχνική πλευρά, αν τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρόταση τη Κομισιόν, αυτό θα ισχύσει. Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε. Και για τους προμηθευτές η επεξεργασία δεδομένων μήπως μετεγκατασταθεί, μήπως μεταφερθεί σε άλλες περιοχές και δεν προστατευτούν τελικά επιχείρησεις στην Ευρώπη. Θέλει κανείς άλλος να κάνει κάποια ερώτηση στους εισηγητές. Η Κομισιό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Απλώς ήθελα να σας πω ότι οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή σας κινείται πάρα πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό και η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει την γραφειοκρατία. Δεν συμφωνούμε όμως με τις ε, με τα όσα ελέγχθηκαν σε αυτή την ενημέρωση ad hoc. Ε, ε, αυτό δεν αφορά τα προφι, δημιουργία προφίλ ή την α, βιβλιογραφία, τα, τη συλλογή, αν θέλει, τη συγκέντρωση ε, εγγράφων ε, ή την μετακίνηση σε τρίτες χώρες. Το profiling επιτρέπεται αλλά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που εφαρμόζονται. Και δεν υπάρχει καμία διαφορά με την ισχύουσα νομοθεσία ούτως ή άλλως. Επομένως, σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία διαφωνούμε με την ενημέρωση που έγινε. Η πρόταση για την καταχώρηση δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν ε, την λειτουργία τους, αλλά θα πρέπει να ε, δούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις και θα πρέπει να ε, δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Η συνάδελφος Άντερς Εξετάζοντας αυτή την έκθεση είδα ότι τα περισσότερα από τα μοντέλα της ε, αγοράς αναλύονται από μερικανικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Μήπως θα μπορούσατε να ε, μας πείτε λίγο για τους ε, ευρωπαίους, ευρωπαϊκούς φορείς τέλος πάντων. Ο τομέας αυτός φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρος, αλλά δεν έχετε μπει σε πολλές λεπτομέρειες. Μήπως θα μπορούσατε για την, για την προστασία των δεδομένων να, και τη βελτίωσή τους να μιλήσετε λίγο παραπάνω για τι γίνεται από τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, έχετε τρία λεπτά ο καθένας για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τουλάχιστον τα δύο πρώτα ερωτήματα για το πώς επηρεάζει κυρίως το άρθρο 20 τα περί profiling. Αυτό το οποίο μάθαμε μετά από συνεντέξεις που είχαμε με διαφόρους και από ήπα και από Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορες δεξιότητες και διάφορες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μικρές και μεγάλες, φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νεοειδριόμενες μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το profiling. Και λόγω της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις και αναπτύσσουν και τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε καινοτόμα συστήματα για ανώνυμα προφίλ. και προσπαθούν να τηρήσουν τις διατάξεις οδηγίας για την προστασία των δεδομένων ε, με, διάφορες, ε, με διάφορους τρόπους. Όμως αυτές ε, δεν τις δέχεται ο νέος κανονισμός. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αν μιλάμε για ομαδικό ή για ατομικό προφίλ και αν μπορεί να έχουμε ανωνυμοποίηση ή όχι. Έχουμε το, την, άμεσο marketing και την άμεση διαφήμιση και το profiling επίσης. Έχουμε και το άρθρο 19, τμήμα 2 του κανονισμού. Επίσης, που έχει ε, μεταξύ άλλων ε, μία διάταξη για το δικαίωμα ένστασης. Άρα πρέπει να δούμε και τα άλλα άρθρα, ε, τα συναφή προς το άρθρο 20 που επηρεάζουν επίσης. Το συμπέρασμα βέβαια είναι ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση και γι' αυτό άλλωστε κάναμε και αυτή τη σύσταση. Να υπάρξει διάκριση λοιπόν μεταξύ των ανώνυμων ομαδικών προφίλ που δεν επηρεάζουν τα προσωπικά δεδομένα και τα μη ανώνυμα δεδομένα που μπορούν να συνδεθούν με τα καταχωρισμένα πρόσωπα αυτά τα data subjects. Και έχουμε τη σχετική οδηγία του 90. Αυτές οι δύο μορφές πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς. Αυτή θα πρέπει να είναι διάξει από την οδηγία του 95. Ο κύριος Κέιβ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που πάρνω, βέβαια και να προσθέσω ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πράγματι τη θέση τους την επηρεάζουν διάφορα πράγματα, όπως εάν αυτές που έχουν μια μικρή βάση πελατών και λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν κάποιες ώρες δεν μπορούν να, δίνουν, ε, να εξασφαλίζουν τα υψηλά επίπεδα συγκατάθεσης για να μπορούν να προστατεύουν ε, την ε, τα προσωπικά δεδομένα μέσα στα επιχειρηματικά τους μοντέλ. Αυτό το είδαμε ε, και με μεγάλα με τις μεγάλες επιχειρήσεις και στις ήπα. Κάποιοι επιλέγουν προφίλ διαφορετικά από τις προτιμήσεις τους στο Facebook, παραδείγματος χάρη. Άρα το θέμα δεν είναι αν κάποιο μπορεί να συμμορφωθεί ή όχι. Τελικά. Πώ μπορεί να εξασφαλιστεί όμω η νομική συμμόρφωση για να μπορεί κανεί να ε, δραστηριοποιείται στην αγορά. Εκεί βλέπουμε οι μικρέ επιχειρήσει να υπολείπονται των μεγαλύτερων που έχουν λιγότερες δυσκολίες. Και θα πρέπει και να δούμε και τις ε, υπηρεσίες που σχετίζονται. Πρέπει οι ευθύνε που αναλαμβάνονται, οι υποχρεώσει που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσει να μπορούν να τι ελέγχουν. Γιατί το θέμα δεν είναι αν, υπάρχουν, είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά, αλλά αν η αγορά μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να εντοπίσει τη σωστή προστασία των προσωπικών δεδομένων και να τη διαθέσει. Η ΜΜΕ που είναι και επεξεργαστέ πλέον δεδομένων, καταλαβαίνουμε αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα. Βγάλουν πέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα βάρη τα οποία αναλαμβάνουν. Πώς θα τους δώσουμε δε απαραίτητα, τα απαραίτητα κίνητρα για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των καταχωρισμένων προσώπων. Έχουμε και τους ελεκτές δεδομένων που ε, συλλέγουν τα δεδομένα. Και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και για τις βασικές υπηρεσίες λοιπόν και για την ε, προστασία προσωπικών δεδομένων έχουμε δύο αγορές και το θέμα να λειτουργούν και δύο σωστά και να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Uh, σε ό,τι αφορά και κάποια παρατήρηση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, πράγματι είναι σωστό αυτό ότι την παροχή υπηρεσιών ε, την, ε, στην αγορά υπηρεσιών. Μάλλον κυριαρχούν μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις. Βέβαια δεν θα πρέπει να δούμε μόνο το θέμα αυτό ε, υπό το κατά πόσον ε, προστατεύουν ε, τα προσωπικά δεμένα ή όχι, γιατί έχουν να προστατεύσουν και τα συμφέροντα των πελατών τους. Κάναμε πολλές συνεντεύξεις και πολλοί μας επισήμαναν τα εμπόδια που υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά είδαμε ότι είναι και πολιτικού χαρακτήρα αλλά και σχετίζονται και με την αγορά πολλές φορές οι ενστάσεις. Θα μπορούσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις να βρούμε τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την προστασία της προσωπικής ζωής. Δεν υπάρχουν ε, μόνο στην Ευρώπη αλλά και στη ΣΥΠΑ πολύ καλά παραδείγματα ανωνυμοποίησης. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα τέλος πάντων να ευχαριστήσουμε τους δύο προσκεκλημένους μας για την ε, συνεισφορά τους και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε τον Υπουργό Σιλικιώτη, τον κύριο Σιλικιώτη, Bene, ringraziamo il Ministro Sirichiotis per la sua presenza, Ministro del Commercio, dell'Industria, del Turismo, della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea che που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποδεχτεί την πρόσκλησή μας για να δούμε τα πορίσματα του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας μαζί και να κάνουμε μια συζήτηση και για το τι επίκειται το επόμενο εξάμεινο. Να, δούμε, να δώσω το λόγο στον Υπουργό για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ ε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Αντιπρόεδρε και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίντρε, κυρίες και κύριοι. Όταν τον περασμένο Ιούλιο αναλάβαμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας παρουσίασα τις βασικές μας προτεραιότητες και τα θέματα που καλούμασταν να διαχειριστούμε, όπως αυτά είχαν καθοριστεί μέσα στο πλαίσιο του τρίου της Προεδρίας Δανία-Κύπρος. Σήμερα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εξάμεινη θητεία της Κυπριακής Προεδρίας, επανέρχομαι για να σας παρουσιάσω τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας. Η σημερινή συνοπτική παρουσίαση του έργου που επιτελέσαμε κατά τη διάρκεια της εξάμεινης ιδείας μας έχει συνεπώς μια διάσταση λογοδοσίας της Προεδρίας του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα όμως εξυπηρετεί και μια αναγκαιότητα, ότι δηλαδή στη δράση και στις πολιτικές που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό σκηνικό που εξακολουθεί να υπάρχει και να μας ταλαιπωρεί στην Ευρώπη, η πρόθεση δράσεων και πολιτικών που θα μας βγάζουν από την ύφεση, θα τονώσουν την ανάπτυξη και θα επενεργήσουν θετικά στην ανάκαψη της οικονομίας μας, αποτελεί το ζητούμενο. Στην Επιτροπή σας υπάρχουν κάποιοι σημαντικότατοι πυλώνες πολιτικής, όπως η βιομηχανία, η έρευνα και η ενέργεια, που μπορούν να αποτελέσουν τους καταλήτες για την αντιστροφή του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος. Επικεντρώνοντας την παρουσίασή μου στα θέματα της αρμοδιότητας μου, τη βιομηχανία και την ενέργεια, σας διαβεβαιώ ότι η Κυπριακή Προεδρία τους τελευταίους έξι μήνες εργάστηκε έντιμα, με συνέπεια και ακούραστα για μια καλύτερη και πιο αλληλέγγυα Ευρώπη, πρώτα και κύρια για τους πολίτες της. Για μια Ευρώπη που θα ξαναβρει το δρόμο της προς την ευημερία, την ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο των εργασιών δύο συμβουλίων ανταγωνιστικότητα, η Κυπριακή Προεδρία πρόθεσε συμπεράσματα σε κέριου τομεί για την πρόθεση της καινοτομία και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και για την τόνωση τη ανάπτυξη και απασχόληση και συνεπώ τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα κράτη μας. Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα τη 11η Οκτωβρίου υιοθέτησε ομόφωνα το Συμβούλιο κείμενων πολιτικών συμπερασμάτων για τι βασικέ τεχνολογίε γενική εφαρμογή. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία των τεχνολογιών αυτών ανήκουν η μικρο- τα προηγμένα υλικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, η φωτονική, η νανοτεχνολογία και τα ευφύ συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Στην παρούσα φάση η Ευρώπη διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο και στις έξι επιμέρους τεχνολογίας διατηρώντας ένα ποσοστό περίπου 32% στις σχετικές αιτήσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί από το 1991 ως το 2008. Εν τούτης, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που, που αξιοποιούνται εμπορικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά από την Κίνα και την Κορέα. Γενικά η Ευρώπη δεν καταφέρνει να κεφαλοποιεί πλήρως τη γνώση που παράγεται και να μετατρέπει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα και υπηρεσίες. Με αυτήν την αναφορά μου δίνεται ευκαιρία παρεθετικά να εκφράσω την ικανοποίηση μου από το γεγονός ότι μετά από τέσσερις δεκαετίες καταλήξαμε στη συμφωνία στη δέσμη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους έξι μήνες εργαστήκαμε πολύ σκληρά σε αυτό το φάκελο και δεν μπορώ παρά να νιώθω ιδιαίτερη τιμή που η Κυπριακή Προεδρία κλείδωσε αυτή τη συμφωνία αναγνωρίζοντα ταυτόχρονα την τεράστια συμβολή προηγούμενων προεδριών αλλά και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτήν τη θετική κατάληξη. Για να επανέλθω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, να προσθέσω πως σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήθηκε και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη καινοτομία για τις πρώτες ύλε και δρομολογήθηκε η ανάπτυξη του σχετικού σταδικού σχεδίου δράσης. Η συγκεκριμένη σύμπραξη στοχεύει σε μη ενεργειακές, μη γεωργικές πρωτεσίλες που θα συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε αυτό, τον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινό στόχο τη συγκεκριμένη σύμπραξη καινοτομία είναι να πραγματοποιήσει η Ευρώπη ω το 2020 ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της εξάρτησής της από την εισαγωγή πρώτων υλών. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Αντεγωνιστικότητα της 10 η Δεκεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υιοθέτησε ομόφωνα κείμενο πολιτικών συμπερασμάτων για την ανασκόπηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα τέσσερα πέπτα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ το 80% των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και ανάπτυξη προέρχεται από τη βιομηχανική παραγωγή. Στο κείμενο των συμπερασμάτων επισημαίνεται ότι ο ρόλος της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό την επίδευξη βιώσιμης ανάπτυξη, τη δημιουργία υψηλή αξία, απασχόληση και την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η ανάληψη άμεση δράση θα πρέπει να συμβάλλει σε αναστροφή τη σημερινή ηφαισιακής τάση, αυξάνοντα το μερίδιο τη βιομηχανία στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τρέχον επίπεδο του 16,5% ως το 20% το 2020 σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτέλεσε μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και τέθηκε στην ατζέντα του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στην Κύπρο. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στην ανάγκη για προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας ως βασικούς πυλώνες για την επιστροφή της Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη. Οι τρόποι στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να οδηγηθούν στην ανάπτυξη συζητήθηκαν ακόμη την πρώτη συνέλευση για τα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία στις 15-16 Νοεμβρίου. Οι συζητήσεις που διεξήχθηκαν κατέδειξαν ότι Όπω και οι προτεραιότητε της ευρωπαϊκή πράξη για τι Μικρομεσαίες επιχειρήσει, γνωστή ως Small Business Act, τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσει στην Ευρώπη είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε άλλε άγορε, κυρίως εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η μείωση του διοικητικού άχθου. Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχρήσεις 2014-2020, θα ήθελα να συνημερώσω ότι παρά τη βούληση της Κυπριακής Προεδρίας να επιταχύνουμε τη διαδικασία, οι δυο διαδοχικέ αναβολές της ψηφοφορίας στην Επιτροπή σας μας απέτρεψαν από το να προχωρήσουμε σε τριλόγους και να έχουμε μία συμφωνία. Στον τομέα της ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει. Συγκεκριμένα, επιτύχαμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά στην πρόταση κανονισμού για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, υιοθετήθηκα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος επί της προτινόμενης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια στις υπεράχτιε δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και ολοκληρώθηκε η διαδικασία υιοθέτηση του κανονισμού για τη σύμμαση του εξοπλισμού γραφείου Energy Star, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του 20% ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοργανώσεων επιτυχία στην Κύπρο, υπουργική διάσκεψη μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών τη Νοτιοανατολική Μεσογείου με αντικείμενο τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασία στα θέματα ασφάλεια, τη υπεράκτητες δραστηριότητες αλλά και τη ενίσχυση τη ασφάλεια και του ενεργειακού εφοδιασμού. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι, όπω γνωρίζετε, και από την παρουσίαση που είχα κάνει στην Επιτροπή σα με την αλέψη τη Προεδρία τον περασμένο Ιούλιο, η επίδεξη συμφωνία επί της πρόταση κανονισμού για τι ενεργειακέ υποδομέ αποτελούσε την πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να εκφράσω τι θερμέ μου ευχαριστίες για τη σημαντικότητα τη συμβολή σα και την άψογη συνεργασία που είχαμε τόσο μαζί σα, κυρία Πρόεδρε όσο και τα μέλη τη επιτροπή σα και ειδικότερα με τον εισηγητή τον κύριο Αντώνιο Κορέρα Τεκάμπος με αποτέλεσμα την ευτυχή αυτή κατάληξη του εν λόγω φακέλου. Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο γιατί θα επιτρέψει την έγκαιρη επιλογή των έργων κοινού ενδιαφέροντος και τη σύνταξη της πρώτης πανευρωπαϊκής λίστας εντός του 2013, αλλά κυρίως γιατί ο κανονισμός αυτός είναι κέριος για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης αφού θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη, στην τόνωση της απασχόλησης και στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας που αφορούν στο σύνολο της Ένωσης είναι ζωτική σημασίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014, καθώς επίσης και για την άρση της απομόνωσης όλων των κρατών μελών μέχρι το 2015, θα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων μας για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2020, ενώ θα βοηθήσει στην προετοιμασία των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης για τον μακροχρόνιο ορίζοντα του 2050. Η επιτυχία αυτή επί της πρώτας κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομίες αποτελεί άλλη μια απόδειξη του πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε όταν υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί την κοινή μας απάντηση και συνεισφορά προς την Ένωση για έξοδο από την υφιστάμενη δύσκολη οικονομική κρίση που διανύουμε κατά τη δύσκολη παρούσα οικονομική συγκυρία. Μια άλλη βασική μα προτεραιότητα αποτέλεσε η υιοθέτηση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στι 3 Δεκεμβρίου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τα συμπεράσματα στηρίχθηκαν στη σχετική ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώ επίση στι θέσει των κρατών μελών όπω αυτέ εκφράστηκαν στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας που προγραμματοποιήθηκε στη Λευκοσία στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως βεβαίως και στις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, όπως εκφράστηκαν από μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα από τον εισηγητή του θέματος, τον κύριο Τούρμες, που ήταν παρόν στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας που προγραμματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Στο κείμενο των συμπερασμάτων δίδεται ιδιαίτερη έφαση στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην καλύτερη σωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά, στη συνεργασία και στην ενίσχυση της εμπορίας των ΑΠΕ μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και με τρίτες χώρες, στην ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών, στην προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, ενωτώθηκαν και οι βάσεις για τη μελλοντική δράση μετά το 2020 προς την κατεύθυνση της στήριξης των ανώσιμων πηγών ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παράγεται μέσω υπεράχτιων δραστηριοτήτων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διαμόρφωση ενός σωστού νομικού πλαισίου που θα μας βοηθά στην άμεση αντιμετώπιση τυχών μεγάλων ατυχημάτων με απρόβλεπτες συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητας δραστηριότητες υδρογοναθράκων τέθηκε πολύ ψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας και αποτέλεσε μια ακόμα βασική μας προτεραιότητα. Αρχικά εργαστήκαμε εντατικά και συστηματικά για την ομαλή μετατροπή της νομικής βάσης της εν λόγω πρότασης της Επιτροπής από κανονισμό σε οδηγία και τελικά πετύχαμε ουσιαστική πρόοδο εντός του Συμβουλίου με αποτέλεσμα να λάβουμε την απαραίτητη διαπραγματευτική εντολή για την επίσημη έναξη των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή σας. Ο πρώτος τρίλογος που πραγματοποιήσαμε το τέλος του προηγούμενου μήνα με τα μέλη της Επιτροπής σας και ειδικότερα τον εισηγητή τον κύριο, τον κύριο Μπέλετ δημιουργεί ένα σημαντικό momentum και θέτει τις βάσεις για την επίδευξη μιας ταχείας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση κατά το επόμενο τρίμηνο. Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει να διατηρηθεί και όλα τα μέρη να συνεχίσουν με την ίδια ένταση τις εργασίες τους και είμαι βέβαιος ότι δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά από την επίδευξη συμφωνίας. Η προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της υπεράκτιας ασφάλειας δεν σταμάτησε εδώ. Στι 13 Δεκεμβρίου η Κυπριακή Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώσαμε στην Κύπρο υπουργική διάσκεψη μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των χωρών τη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο της συνεργασία στον τομέα της ενέργεια. Βασικά θέματα συζήτηση αποτέλεσαν η ασφάλεια στις υπεράχτης δραστηριότητες υδρογοναθράκων, και ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού από και προς την Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσω της πιθανής δημιουργίας του Νοτιοανατολικού Μεσογειακού Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη υιοθέτηση από τις συμμετέχοντες κοινή διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τους προσανατολισμούς μας στα θέματα αυτά. Η θάλασσα δεν γνωρίζει σύνορα. Οπότε και δεν αρκεί μόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης να εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ιδιότερα όταν σε εμίκλειστες θάλασσες, όπως η Μεσόγειος, όπου οι γειτονικέ μας τρίτες χώρες, μετά από τις πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περιοχή, ολοένα και εντείνουν τις υπεράκτιες τους δραστηριότητες για τον λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητη την ενίσχυση της συνεργασίας και την πρόθεση των ύψιστων προτύπων ασφάλειας όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και με τις τρίτες γειτονικές μας χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη που έδωσαν τον παρόν τους στη συνάντηση στη Λευκοσία. Είμαι βέβαιος ότι όπως όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε το να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου αυτέ τι χώρε δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όμω το γεγονό ότι η Κύπρο ήταν και παραμείνει ένα έντιμο φίλο και συνεργάτη με όλου του γειτονέ τη, αλλά και επίδη επικοινωνία τη Νοτιοανατολική Μεσογείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία αυτή τη υπουργική συνάντηση. Μεταφέροντα το θέμα τη ασφάλεια στι υπεράκτιε δραστηριότητε σε γενικότερο πλαίσιο, Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε τη δυνατότητα ως Ένωση και θα πρέπει να επιδιώξουμε να λάβουμε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και πρόθεση σε παγκόσμιο επίπεδο υψηλών προτύπων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις υπεράκτητες δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία αποτελεί κατά νόψη μας το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να πω ότι και η συνάντηση αυτού του εξαμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετροπαραγωγικό Χωρό, είχε ως αντικείμενο την ασφάλεια ε, στις υπεράκτιες ε, εξορίξεις. Παράλληλα, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 3 Δεκεμβρίου, η Προεδρία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία αποτελείται από έξι τομείς πολιτικής την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εσωτερική αγορά ενέργειας και τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις υποδομές, τις διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια. Τέλος, ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, υιοθετήθηκε απόφαση Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 10ο Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου στο Μαυροβούνιο, απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μόνιμο Συμβούλιο Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 12 Δεκεμβρίου, καθώς και απόφαση του Συμβουλίου για επέκταση του χρονοδιαγράμματο εφαρμογής από τη Μολδαβία του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009 κάθετος 73 της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2020. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην επερχόμενη Ελλαδική Προεδρία και να διαβιώσω τον Ιρλανδό ομολογό μου ότι θα είμαστε δίπλα τους για να στηρίξουμε το έργο του. Πριν όμως να ολοκληρώσω θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου Πρώτα-πρώτα στην Επιτροπή και τους αρμόδιους επίτροπους, τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη και τον Επίτροπο Νότιγκερ, στα κράτη-μέλη που μέσα από τη ε, συμβολή τους βοήθησαν στο να ολοκληρώσουμε τους φακέλους, την Επιτροπή, την Πρόεδρο της ε, Κυριευτικής Επιτροπής Ίντρε και τα μέλη της Επιτροπής, σας δηλαδή, αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου, τους λειτουργούς των Κωνσταντίνων Καραγιώργη, το Γιώργο Καμπανταϊδάκη, το Χρήστο Κογάκη, τη Λεωνή Θεοδωρίδου, τον Αναστάσιο Παπανδρέου και πολλούς άλλους λειτουργούς που όλον αυτό το εξάμενο δούλεψαν ακούραστα και με συνέπεια για να διεκπαιρωθεί αυτός ο μεγάλος όγκος δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό τον κύριο Σιλικιώτη για τη διεξοδική αυτή, λεπτομερέστατη και ακριβέστατη παρουσίαση. Τώρα, στα πλαίσια της συζήτησης έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τούρμες. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, είναι κρίμα να είναι τόσοι λίγοι βουλευτές ε, παρόντες στην αίθουσα. Δεν θα πρέπει όμως να το δείτε προσωπικά. Εδώ ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος ασχολήθηκε σε μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, το ίδιο και εγώ, Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το πώ εξελίχθηκε αυτό το τελευταίο εξάμεινο, παρά τις δυσκολίες, τις οικονομικέ που αντιμετωπίζει η χώρα σας δεδομένων των ε, πιέσεων, των εντάσεων στην ε, Συρία, το Λίβανο, στην άμεση γειτονία σα, ε, παρόλε αυτέ τι δυσκολίε, εσεί και οι συνεργάτε σα επικεντρωθήκατε με μεγάλη επιτυχία στι ενεργειακέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Κορέιντε Κάμπο επικεντρώθηκε στις ενεργειακές υποδομές. Εγώ πάλι ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω για, το, για την εξαιρετική περάτωση του θέματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. ο στόχος που έχει τεθεί, η ανανέωση των εθνικών συστημάτων και η ενίσχυσή τους ε, με την συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ ε, σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Με την επίσκεψή μας στην Κύπρο ήταν ε, μεγάλη ικανοποίηση να δούμε ότι προχώρησαν τα σχέδια για την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια και για περαιτέρω προγράμματα, καθώς και την ε, χρήση του θαλασσινού, την αξιοποίηση του θαλασσινού νερού. Είναι πολύ καλό να προωθηθούν όλες αυτές οι νέες ιδέες στην λεκάνη της Μεσογείου. Και στην όλη εξέταση του θέματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σημαντικό ότι προωθήθηκε και το σύστημα για την ανταλλαγή δικαιωμάτων ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά είναι καθοριστική σημασία για να διασφαλίσουμε, για να εξασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν είναι υπέρ αυτού του συστήματος εμπορίας Και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι του ΕΛΚ που δεν θέλουν το σύστημα αυτό να ισχύει ως έχει. Όμως το Συμβούλιο πολύ σωστά είπε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστική σημασία η ισχύ του συστήματος αυτού. Είναι πολύ σημαντικά επίση όσο αναφέρονται στο έγγραφο για τις ε, κλιματικέ αλλαγέ. Και ήθελε εδώ για την τελευταία Υπουργική Σύνοδο να σας ρωτήσω πώς έχουν εξελίξει σε σχέση με την εσωτερική αγορά και την προσέγγιση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η γενική αίσθηση που, που επικράτησε μετά τη συνάντηση αυτή πριν από δύο εβδομάδες. διότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε την ε, εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά για την ενέργεια. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην κατάσταση τη δεκαετία του 80 όπω την εσωτερική αυτή αγορά προφανώ. Γι' αυτό περιμένουμε την άποψή σα. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε ο κύριο Κορέα Τεκάμπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριο Ηλικιώτης, ήταν χαρά μας ε, που ήρθαν εδώ σήμερα και τον ακούσαμε σε όσα μας είπε. να τον ευχαριστήσω λοιπόν πάνω απ' όλα και να συγχαρώ την Κυπριακή Προεδρία για το αποτέλεσμα των προτεραιοτήτων που έθεσε και στα πλαίσια των εργασιών της δικής μας Επιτροπής. Νομίζω ότι η έγκριση του Ευρωπαϊκού Διπλώματο ευρεσιτεχνία, ε, οι ενεργειακές υποδομέ, ε, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και η σύνοδος, η περιφερειακή σύνοδος για την ενέργεια θα παραμένουν στην ιστορία τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Απλώς να πω το εξή. Ολοκληρώθηκε το εξάμεινο της Προεδρίας από μια χώρα που βρίσκεται στην νότια περιφέρεια της Ευρώπης. και όμως κατάφερε να συντονίσει αμφιλεγόμενες απόψεις και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας ένα αίσιο πέρας. Κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα, Η συνεργασία με τον πρέσβη Ζωδιάτη και κυρίως ε, και τους υπόλοιπου συνεργάτες του ήταν υποδειγματική. Ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ήταν θεμελιώδη, διότι ακριβώς διευκόλυνε τις συνομιλίες μεταξύ των δύο υπεύθυνων νομοθετών, ε, όσων είναι αρμόδιοι για την συναπόφαση δηλαδή διευκολύνθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ τους και μπορέσαμε να επεξεργαστούμε βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Μετά την έγκριση του κανονισμού αυτού, η Ευρώπη θα αποκτήσει πλέον μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά που δεν έχει ακόμη. Δεν την διαθέτει. Θα μπορέσει πλέον να τη δημιουργήσει. Θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα λεγόμενα bottlenecks και τις ενεργειακές ε, δυσχέρειες που έχουμε αντιμετωπίσει ως τώρα. Και η δική σας ε, χώρα τις έχει γνωρίσει και άλλες χώρες, όπως η δική μου ή οι χώρες της Βαλτικής. Η άρση των φραγμών σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ενέργειας. Είναι αδιανόητο μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία το 2020 να αποφασίζει να πάψει την πυρηνική της παραγωγή αλλά δεν μπορεί να κλείνει τις πόρτες της στην ενέργεια που έρχεται από τον Νότο. και να αποφασίζει να εξαρτηθεί πλήρω από την αιωλική ενέργεια, από το αέριο που εισάγεται από την Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει καμία λογική κάτι τέτοιο. Εάν κλείσουμε τις πύλες ε, από τον Νότο, η Γερμανία αναγκαστικά θα στρεφόταν προς το Βορρά. Δεν χρειάζεται να παραμείνουν μόνον αυτοί οι διάβλοι. Χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς. Μηχανισμούς για τον συντονισμό των ενεργειακών δικτύων, κάτι που δεν υπήρχε ακόμη. Το χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε τις απότομες ε, ελλείψεις ε, στην ενέργεια, τις απότομες διακοπές και τα blackout. Και πάλι, Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, να σας συγχαρώ για την Σύνοδο για την Ενέργεια και την κυρία Σαρτόρη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε μια δύσκολη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Καταφέραμε να αποσπάσουμε ένα έσω αποτέλεσμα, χάρη όμως και στις προσπάθειες ε, και τις διπλωματικές ικανότητες του κ. Ζωδιάτη και όλη της, της του, του Γενικού Διευθυντή, του Ευρωπαίου Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένο με τα θέματα ενέργεια, που καταφέραμε να, ε, με τον οποίο καταφέραμε να έχουμε μια άριστη συνεργασία. Σα ευχαριστώ όλου και εσά ιδίω, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Μετά από τι παρεμβάσει αυτέ, για την ολοκλήρωση τη συνάντησή μα, να δώσω το λόγο και πάλι στον ε, Υπουργό εάν θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ήθελα να, ε, καταρχήν να ευχαριστήσω ε, και τον κύριο Τούρμες και τον κύριο Κορέλια Τεκάμπος η οποία η συνεργασία μαζί τους ε, θα έλεγα ήταν άψογη και υποδειγματική. Να πω ότι ε, βεβαίως όταν αναφερόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κύριε Τούρμη αυτό που συζητήσαμε και στη Σύνοδο στην Κύπρο αλλά και στο Συμβούλιο η, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει την πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα που έχει ε, διεθνώς. Ε, πέρα δηλαδή από την κάλυψη των δικών της ε, αναγκών και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, θα πρέπει ακριβώς να συνεχίσει αυτή την πορεία και θεωρώ ότι τα συμπεράσματα της 3 Δεκεμβρίου είναι μια ισχυρή πολιτική βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική της για τις ανάλυσιμες πηγές ενέργειας στην πορεία προς το 2050. Ε, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν μιλούμε για εσωτερική αγορά μετά από τη συζήτηση και στις 3 του Δεκέμβρη με την ενημέρωση της έκθεσης ε, προώρου και για αυτόν τον τομέα επαναλήφθηκε η ισχυρή δέσμευση που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι ε, μέχρι το 2014 πρέπει να ελοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ε, και εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε με πολύ συνέπεια και θα έλεγα αποφασιστικότητα την ανάγκη για ελοποίηση αυτού του στόχου και θεωρώ πολύ σημαντικό, το ανάφερε και ο κύριος ε, Κάμπος, ότι συμφωνία, η κατάληξη για την υλοποίηση του κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομές θα βοηθήσει ακριβώς ε, για να ονοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας. Ε, και έχετε ε, δίκιο κύριε Κάμπος όταν αναφέρεστε ε, στην ανάγκη να υπάρξει η σύνδεση στην Ευρώπη. Ε, σε διάφορες περιοχές υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να έβρουμε τον τρόπο να υπάρξει αυτή η αλληλουχία και συνεργασία γιατί τα θέματα α, της εσωτερικής ασφάλειας, η άσκηση της απομόνωσης των κρατών μελών, η ενίσχυση των διευρωπαϊκών υποδομών θα βοηθήσει πρώτα και κύρια να αποκτήσει ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα είναι προ όφελο και των πολιτών, των καταναλωτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Αλλά θα ήθελα να κάνω ε, μια προέκταση, να δώσω ακόμα μια διαστασή. Η, η συζήτηση που έγινε στην Κύπρο και η ανάγκη για να συνδεθεί η Κύπρος με την περιοχή της Νοτανατολικής Μεσογείου και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πίτροπος ε, Ότιγκερ στη Σύνοδο στην Κύπρο έχει αναφέρει ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία ε, στην ενεργειακή τροφοδοσία από τη βορρά, από τη βόρεια θάλασσα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Μεσογείου είναι μια ισχυρή βάση για να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και ιδιαίτερα η ενεργειακή ασφάλεια των νότιων κρατών μελών, των μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως και στη Σύνοδο στη Λευκοσία θέσαμε ακόμα μια άλλη Την ανάπτυξη το σχέδιο με, τις νότιες, ε, με τους νότιες γείτονες μας. Και αναφέρομαι στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και στον τομέα των ονάσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να διευρύνουμε από τη μια να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά αλλά να διευρύνουμε την αγορά ενέργειας στην Ευρώπη σε συνεργασία όχι μόνο με, τις, ε, με τους ανατολικούς γειτονές μας αλλά και με τους νότιους γειτονές μας ε, και εδώ θα συμβάλλουν πολύ αποφασιστικά ε, τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και οι ενεργειακές υποδομές. Ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στη δουλειά μας. Ε, έχετε δίκιο κύριε Γκάμπος, που αναφερθήκετε και στο, ίσως ήταν μια παράληψή μου, στον πρέσβη τον Γιώργο τον η οποία η παρουσία του ως Προεδρεύον της Κορομπέρ και στο συντονισμό των συνεργατών μας εδώ στις Βρυξέλλες ήταν αποφασιστική για να προωθούν αυτοί οι φακέλοι. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Σαστορή, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω για τη στενή και αποδοτική συνεργασία μας όλων αυτών το εξάμεινο να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σας εργασίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε όλους για το έργο σας. Bene, proseguiamo. Ωραία. Ας ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας, καλωσορίζοντας την κυρία Ελένη Μαύρου, ε, η οποία είναι υπουργό Εσωτερικών, αλλά στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και, περιλαμβάνονται και τα θέματα της έρευνας. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δική της ομιλία, την ομιλία της κυρίας Μαύρου για τα αποτελέσματα του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Good day, everybody. I understand you have a busy... Καλημέρα σε όλε και όλου. Ξέρω ότι είναι αρκετά βεβαρημένη η ημερήσια διάταξη. Θα προσπαθήσω να είμαι στον πιο σύντομη και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να συνεχίσω στα ελληνικά. Ε, κυρία μέλη του, αγαπητή, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, καταρχάς επιτρέψτε μου να σα ευχαριστήσω εσά προσωπικά κυρία Πρόεδρε καθώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Αναλάβαμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Με την οικονομική κρίση να ταλανίζει την Ευρώπη και να ταρακουνά τα θεμέλια και τις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έχει τονιστεί πολλές φορές ότι ο τρόπος εξόδου από την κρίση είναι η ενδυνάμωση πολιτικών ανάπτυξης και κυρίως η πρόθεση επενδύσεων και μέτρων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Γι' αυτό και η χρονική περίοδος που πήραμε τη σκητάλη από την Δανική Προεδρία, ειδικά για τα αναπτυξιακά αυτά θέματα, είναι σημαδιακή αφού εκτός από την οικονομική κρίση η περίοδος αυτή συνέπιπτε με τη διαπραγμάτευση του επόμενου προγράμματος πλαισίου για έρευνα και καινοτομία του Ορίζοντα 2020. Όπως γνωρίζετε, ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί το πρόγραμμα αναβαρχίδα της Ένωσης σε θέματα έρευνας και καινοτομίας για την επόμενη επιθετία και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα αποτελέσει ένα εργαλείο έξυπνης χρηματοδότησης της Ένωσης στις κατάλληλες ερευνητικές προτεραιότητες ε, και θα συμβάλλει στην έξοδο της Ένωσης από την οικονομική κρίση το συντομότερο δυνατό. Ε, σας είχε ενημερώσει ο προκάτοχος μου, ο κύριος Σταύρος Μαλάς, τον περασμένο Ιούλιο για τους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η Κυπριακή Προεδρία και τις προτεραιότητες της στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Θα ήθελα να αρχίσω την ενημέρωση για τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών με το πιο σημαντικό θέμα, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 που θα καθορίσει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα της έρευνας για την επόμενη επταετία μεταξύ 2014 και 2020 για τους ε, κανόνες συμμετοχής στον ορίζοντα 2020. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου έγιναν έντονες συζητήσεις στο Συμβούλιο με τα κύρια πολιτικά θέματα να συζητούνται επίσης μεταξύ των Υπουργών και στο άτυπο Συμβούλιο που έγινε στη Λευκοσία το καλοκαίρι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των κανόνων συμμετοχής ήταν η ανάγκη της απλοποίησης των διαδικασιών έτσι ώστε να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα αποτελεσματικό, απλοποιημένο και προσβάσιμο για τον τελικό χρήστη που είναι ο Ευρωπαίος ερευνητής. Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς στο Συμβούλιο το μοντέλο υπολογισμού της επιστροφής άμεσων και έμμεσων δαπανών του προγράμματος, η μισθή των ερευνητών από νέα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως και η ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα. Μετά από δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις, τελικά τον Οκτώβριο, στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, καταφέραμε να συγκεράσουμε τις διστάμενες απόψεις των κρατών μελών και να επιτύχουμε συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου με την υιοθέτηση μερικής γενικής προσέγγισης. Το πρώτο ε, κύριο χαρακτηριστικό αυτής της συμφωνίας ήταν η επιβεβαίωση των κρατών μελών για ένα απλοποιημένο πρόγραμμα πλαίσιο με ένα μοναδικό μοντέλο επιστροφής των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα, με 100% επιστροφή των άμεσων δαπανών σε ένα ερευνητικό έργο, και οριζόντια 25% επιστροφή στο σύνολο των άμεσων δαπανών για τις έμμεσες δαπάνες. Για τις καινοτόμες δράσεις που είναι κοντά στην αγορά κρατήσαμε την πρόταση της Επιτροπής για ποσοστό 70% επιστροφή των άμεσων δαπανών. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς το ποσοστό επιστροφής άμεσων δαπανών θα είναι πάντοτε στο 100%. Το άλλο κύριο χαρακτηριστικό της συμφωνίας ε, του Οκτωβρίου ήταν η εισαγωγή ενός νέου άρθρου για τους μισθούς του προσωπικού που εργάζεται σε έργα του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Με την ε, προσθήκη που έγινε επιτρέπεται σε οργανισμούς που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα του προγράμματος να δίνουν πρόσθετα κίνητρα σε μορφή φιλοδορήματος στους εμπλεκόμενους ερευνητές και στη συνέχεια αυτή η δαπάνη να καλύπτεται από τον ορίζοντα 2020. Φυσικά για να περιοριστούν οι δαπάνες το ανώτατο όριο του φιλοδορήματος έχει καθοριστεί στις 8.000 ε, ευρώ ε, ετησίως. Ε, αυτό είναι το όριο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αναερευνητή που συμμετέχει με πλήρη απασχόληση στο έργο. Η νέα αυτή πρόνοια εισήχθηκε για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα κάποιων κρατών μελών, των οποίων η συμμετοχή στο εφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι συγκριτικά χαμηλότερη και ζητούσαν αύξηση ε, των κινήτρων αυτών. Θα συνεχίσουμε το άλλο μεγάλο μέρος του νομοθετικού πακέτου ορίζοντας 2020, το ειδικό πρόγραμμα, ε, συνδεδεμένο βεβαίως με τον, κύριο, ε, με τον κυρίως ε, κανονισμό. Ε, γι' αυτό και η προσέγγιση που επιλέξαμε στο Συμβούλιο για το ειδικό πρόγραμμα, κάτι που αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει και στο Κοινοβούλιο, ήταν να ακολουθήσουμε τη Γενική Συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο τον περασμένο Μάη για τον κυρίως κανονισμό του ορίζοντα 2020. Στη μερική γενική προσέγγιση που συμφωνήσαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα ε, στο Συμβούλιο, κρατήσαμε τη βασική δομή του προγράμματος που συμφωνήθηκε για τον κυρίως κανονισμό. Υπενθυμίζω ότι οι δομικές αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής ήταν ο διαχωρισμός της κοινωνικής πρόκλησης σε 2 με τη δημιουργία της νέας κοινωνικής πρόκλησης 7 για ασφαλείς κοινωνίες καθώς και εισαγωγή ενός οριζόντιου κουτιού με διατομεακά θέματα και υποστηρικτικές δράσεις. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στο Συμβούλιο ήταν η επιτροπολογία και η μελλοντική διακυβέρνηση του προγράμματος. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο αντικατοπτρίζουν την επιθυμία των κρατών μελών για περισσότερη εμπλοκή στη διακυβέρνηση του προγράμματος, ακολουθώντας εν μέρη το καθεστώς εφαρμογής του υφιστάμενου 7ου προγράμματος πλαισίου. Τέλος, όπως έγινε και στους κανόνες συμμετοχής, υπήρξαν έντονες συζητήσεις για το θέμα διεύρυνσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα ερευνητικών φορέων από όλη την Ευρώπη στο Συμβούλιο συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του χάσματος έρευνας και καινοτομίας στην κοινωνική πρόκληση 6, τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση περιφερειών με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα. Η τελευταία από τις τέσσερις νομοθετικές προτάσεις του πακέτου ορίζοντας 2020 είναι το πρόγραμμα πλαίσιο Euratom που περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες οι οποίες αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν ε, στον τομέα της πυρηνικής έρευνας για την περίοδο 2004-2018. Στη διάρκεια της ε, Προεδρίας ε, υιοθετήσαμε έκθεση προόδου από το Συμβούλιο όπου ουσιαστικά ευθυγραμμίσαμε το νομοθετικό κείμενο με τη συμφωνία του περασμένου Μαΐου επί του κυρίως κανονισμού του ορίζοντα 2020. Από τις συζητήσεις διαφάνηκε ότι στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πυρηνικής ε, ασφάλειας. Για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας κάναμε επίσης σημαντικά ε, βήματα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όπως γνωρίζετε, έχει προταθεί ως αναπόσπαστο μέρος του ορίζοντα 2020. Στη δική μας Προεδρία το Συμβούλιο έχει φτάσει σε μερική συμφωνία και στις δύο νομοθετικές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας για τη μελλοντική του λειτουργία, ε, δηλαδή την πρόταση τροποποίησης του ιδρυτικού κανονισμού του EIT και την πρόταση για τη στρατηγική ατζέντα καινοτομίας του EIT. Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συμβούλιο ήταν το θέμα της δημιουργίας των μελλοντικών κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας για το 2014 και το 2018. Ως αποτέλεσμα των ε, συζητήσεων μας την περασμένη εβδομάδα στις 11 του Δεκέμβρη είναι η δημιουργία ενός πρώτου κύματος τριών κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας το 2014 στους τρεις θεματικούς τομείς που έχουν προταθεί από την Επιτροπή, δηλαδή στην καινοτομία για μια υγιή ζωή και ενεργογύρανση, στις πρώτες ύλε και στα τρόφιμα για το μέλλον. Για το δεύτερο κύμα, μετά το 2017, το Συμβούλιο επέλεξε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, αφήνοντας ε, την ε, επιλογή στα πλαίσια μιας νέας νομοθετικής διαδικασίας συναπόφασης το 2017 λαμβάνοντας υπόψη και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τυχόν νέες θεματικές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Ε, το τελευταίο εξάμηνο προωθήσαμε με γρήγορους ρυθμούς και τις συζητήσεις για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 95% των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας διεξάγονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ε, η ολοκλήρωση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας θα σημάνει και την απρόσκοπτη κυκλοφορία της γνώσης στην Ένωση, την ευκολία κινητικότητας των ερευνητών και την διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της ε, έρευνας. Για τα πιο πάνω μέτρα έχουν προωθηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, συμπεράσματα Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν ομόφωνα την περασμένη εβδομάδα από τους Υπουργούς. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και οργανισμούς, με βάση τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής προωθήσαμε στο Συμβούλιο μια πιο στρατηγική προσέγγιση της Ένωσης για το θέμα αυτό και στο άτυπο Συμβούλιο Έρευνας τον περασμένο Ιούλιο τέθηκαν οι πολιτικές βάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας της Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες με την πιθανή δημιουργία μιας πρωτοβουλίας με βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης, ειδικά για την Ευρωμεσογειακή Περιφέρεια. Παράλληλα με τις εργασίες της Βρυξέλλες έγιναν και στην Κύπρο διάφορα συνέδρια προεδρίας ε, τα οποία ήταν συμπληρωματικά στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων που θέσαμε. Επιγραμματικά αναφέρω ότι τον Νοέμβριο έγινα στην Κύπρο δύο μεγάλα συνέδρια για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ε, τον περασμένο Οκτώβριο ε, πραγματοποιήθηκε συνέδριο Προεδρίας με θέμα την ανοιχτή καινοτομία στον τομέα της υγείας, ενώ λόγω της σημασίας του θέματος της κινητικότητας των ερευνητών έγινε επίσης ε, συνέδριο με θέμα της δράσης Μαρίας Κολτόσκα Κιουρί. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός ήταν ο απολογισμός των κύριων θεμάτων που ε, διαχειριστήκαμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Έχω ε, ενημερωθεί ότι η Επιτροπή Ήτρε στις 28 του Νιόβρη έχει ψηφίσει τις προτινόμενες τροποποιήσεις της στο νομοθετικό πακέτο του Ορίζοντα 2020 και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, ε Τεχνολογίας ε, κάτι που σημαίνει και την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων ε, μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων της Ένωσης για το θέμα στις αρχές του νέου χρόνου. Ο κύριος μας στόχος από την αρχή της Προεδρίας μας ήταν να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον ορίζοντα και το EIT έτσι ώστε το Συμβούλιο να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2012 τις εσωτερικές του διαδικασίες για το νομοθετικό πακέτο. Όπως έχω αναφέρει πιο πάνω, ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί με τέσσερις μερικές γενικές προσεγγίσεις που μαζί με αυτή που έχει επιτευχθεί από τη Δανική Προεδρία για τον κυρίως κανονισμό του ορίζοντα 2020 δίνουν ουσιαστικά το πράσινο φως στην Ιρλανδική Προεδρία να αρχίσει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχές του χρόνου με στόχο την υιοθέτηση του ορίζοντα 2020 πριν το καλοκαίρι του 2013. Θέλω να ευχηθώ με αυτή την ευκαιρία στην Ιρλανδική Προεδρία ε, κάθε επιτυχία σε αυτό τον σημαντικό τομέα. Ε, είναι σημαντικό να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα όλοι μας και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δουλέψει ε, πολύ σκληρά και είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την έγκαιρη έναρξη των προγραμμάτων του Ορίζοντα 2020 την πρώτη του Γενάρη του 2014. Αυτή η δέσμευση στέλνει και τα κατάλληλα μηνύματα στην ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα που περιμένει με ανυπομονησία την έναρξη του ορίζοντα 2020. Τέλος, επιτρέψτε μου ξανά, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να παρουσιάσουμε το έργο της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα επίπεδα αυτό το τελευταίο εξάμεινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μαύρου, την κυρία Ελένη Μαύρου για την παρουσίασή της, η οποία ήταν τόσο συγκεκριμένη όσον αφορά τις εργασίες ε, του Συμβουλίου το τελευταίο εξάμεινο. Τον λόγο τον έχει ο συνάδελφος Όντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Υπουργό για, την, ε, για το ενδιαφέρον που δείξατε και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Θα είδατε ίσως ε, την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας η οποία, και στο Κοινοβούλιο η οποία αποκλίνει λίγο από την άποψη του Συμβουλίου όσον αφορά την βασική έρευνα και το τι και τι εννοούμε πλησίων της αγοράς, κοντά στην αγορά. Σε σχέση με τον ΠΟΕ, διότι όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κοντά στην αγορά, δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε ε, αυτό το οποίο ισχύει, θεωρείται ότι είναι συμβατό με τους κανόνες ε, του ΠΟΕ ή στο Συμβούλιο θεωρείται ότι αυτό το θέμα των επιδοτήσεων δεν ε, θύχθη. Δεύτερη ερώτηση για την απλούστευση. Εμείς ε, πιστεύουμε, εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι η πρόταση της Κομισιό ε, σεβόταν ε, τα κριτήρια της απλούστευση και ίσως εμείς οι βουλευτές να περιπλέξαμε τα πράγματα. Λοιπόν, στο θέμα της απλούστευσης, ποια είναι, ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στο Συμβούλιο, θα παραμείνετε στις απόψεις της Κομισιόν, που οι, αυτές θα είναι από άποψη του Συμβουλίου ή η, η ψηφοφορια στην, της Επιτροπής μας θα επηρεάσει. Επίσης, ε, για το ποσοστό της ε, επιστροφής, ε, πιστεύω, μάλλον θεωρείται ότι ο, η βιομηχανία χρηματοδοτείται επαρκώς σε σχέση με την ψηφοφορία που είχαμε εμεί στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα παραμείνει στο 100%. Δεν θα ξαναπάρω το λόγο, γι' αυτό ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνησή σας και εσάς προσωπικά για την Προεδρία. Δεν είναι εύκολο να ασκεί κανείς Προεδρία και μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε και δύο λόγια για την Τρόικα. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για την χρησιμότητα της, ε, της Τρόικας. Εσείς ε, που ολοκληρώνετε την, ε, το τρίο τέλος πάντων Πολωνία, Πορτογαλία, Κύπρος, τι έγινε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και λυπάμαι ότι δεν, είσα, δεν είχατε κι εσείς προσκληθεί μαζί με τους ε, τρεις άλλους υπεύθυνους ε, της ε, Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είσαστε παρόντες να πάρετε το, το, το Νόμπελ. Ε, είσαστε κι εσείς ε, συνομοθέτες και λυπάμαι πραγματικά που δεν είστε εκεί, το έχω πει ήδη ε, δημόσια. Πάντως ούτως ή άλλως σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Οντί, ο κύριος Τζόνσον έχει το λόγο. Thank you very much and thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια και για την παρουσίαση της Προεδρίας. Είχα την ευκαιρία να ενταχθώ στην διαπραγματευτική ομάδα μου και όδη ηγητή τη ομάδα Άλντε όταν συζητήσαμε το ορίζοντα 2020 και όπως είπε και ο κύριος Οντί θα πω και εγώ κάποια πράγματα σε σχέση με τη δική μας προσέγγιση στην Επιτροπή Ήτρε. Θα ήθελα δύο σχόλια από εσάς. Το πρώτο, επειδή μιλήσατε για αυτά τα 8.000 ευρώ στις συζητήσεις μας όμως, πώς θα σας το πω, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω την προσέγγιση και γιατί λήφθη αυτή η απόφαση στο Συμβούλιο. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να πω, ότι το πρόγραμμα θα κοστίσει περισσότερο. Στις συζητήσεις που είχαμε εμείς, προετοιμάζοντας το όλο θέμα, ακολουθήσαμε την προσέγγιση να υπάρχει μεγαλύτερη μόχλευση στο Horizon 2020 και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δηλαδή, να μπορούμε με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ε, να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες έρευνας. Ε, έχετε εσείς κάποιες απόψεις πώς μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη μόχλευση. Ένα τρόπο σίγουρα είναι η απλούστευση των κανόνων, αλλά μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να υπάρχει, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερη μόχλευση του ποσού, αν έχετε κάποιο σχόλιο. Και δεύτερον, συζητήσαμε κι εμείς πώς θα μπορούσαμε να έχουμε πιο στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικής συνοχής και περιφερειακών ταμείων αφενός και ορίζοντα 2020 αφετέρου. Ένα παράδειγμα είναι το εξής. Όταν συζητήσαμε τα περίπτωση να χρησιμοποιούν διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής με πιο αποτελεσματικό τρόπο και στο όλο πακέτο του ορίζοντα 2020 νομίζω ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι αυτό, δηλαδή να γίνει αυτό μέσω των δραστηριοτικών, των περιφερειακών ταμείων, να υπάρξει μεγαλύτερη δημιουργία υποδομών, capacity building. Αν έχετε να σχολιάσετε και αυτό, βέβαια θα τα συζητήσουμε και με την επόμενη Προεδρία, το επόμενο εξάμεινο. Το Κοινοβούλιο σίγουρα με το Συμβούλιο θα συζητήσει αυτή την προοπτική της μόχλευσης, παραλαμβάνω, ώστε με τους ίδιους πόρους να μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ πολιτικής συνοχής και ορίζοντα 2020. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για το έργο που εκτέλεσε η Προεδρία σας και νομίζω ήταν πολύ καλό για μας γιατί έχουμε πλέον έχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ τον ε, συνάδελφο κύριο Τζόνσον. Δεν έχω κανέναν άλλον που να ζητάει το λόγο και θα δώσω το λόγο στην ε, Υπουργό για να απαντήσει στις ερωτήσεις και για να ολοκληρώσουμε και την ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ. θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί θεωρώ ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε τους επόμενους μήνες σε ό,τι αφορά ε, την, ε, ε, το να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και σε στόχους και σε διαδικασίες. Ε, έχει δίκιο ο κύριος ε, Οντή ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των στόχων των ερευνητικών και της ε, της ε, αγοράς. Αυτά τα θέματα θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ Ιρλανδικής ε, Προεδρίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα της απλοποίησης που είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό για τα προγράμματα των δημοσιονομικών προοπτικών του 2014-2020 και στην περίπτωση του ορίζοντα 2020 η απλοποίηση περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα. Ε, στο Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβρη δεν υιοθετήθηκε το μοντέλο συνολικού κόστους ε, το οποίο ήθελαν ε, πολλές αντιπροσωπείες επειδή το επιχείρημα της ε, απλοποίησης πραγματικά έπεισε ε, πολλούς. Ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει στη συνέχεια να, στις συζητήσεις μας με το Ευρωκοινοβούλιο να, βρούμε ένα τρόπο, να, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Η απλοποίηση είναι μια πολύ σημαντική πτυχή του προγράμματος Ορίζοντας 2020 είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα όλων εκείνων που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη ε, των στόχων της. Γνωρίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις είναι αφιλεγόμενες και ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει τροποποιήσεις ε, στο μοντέλο χρηματοδότησης. Ε, μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου τον Οκτώβρη στην οποία τα κράτη-μέλη πίστηκαν για το πόσο σημαντικό κομμάτι της απλοποίησης είναι το χρηματοδοτικό μοντέλο είμαστε αισιόδοξοι για την συζήτηση που θα έχουμε να κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοι ε, της Ιρλανδικής Προεδρίας θα το χειριστούν ε, δημιουργικά. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι ε, για να προχωρήσω και στην άλλη παρατήρηση ε, του κυρίου Γιώχανσον για τα, για τα κίνητρα τα οποία δίνονται μέσω των κανόνων συμμετοχής στον ορίζοντα 2020. Να διευκρινίσω ότι το Συμβούλιο έκρινε ότι και η απλοποίηση αλλά και αυτή η δυνατότητα να δίνονται πρόσθετες αμοιβέ σχετικά χαμηλού ύψους είναι πολύ σημαντικά τμήματα μιας πολιτικής που θα συμβάλλει θετικά στη διεύρυνση της ε, συμμετοχής. Ε, η Προεδρία θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία ε, στο Συμβούλιο είναι σημαντική Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πιστεί ε, για την αξία της απλοποίησης των ε, διαδικασιών. Ε, οι 8.000 ευρώ ετησίως ανά ερευνητή είναι κίνητρο για τους ερευνητές κυρίως από ε, καινούργια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 2020. Ε, Αν θέλετε είναι μια προσπάθεια να παρεμβάλλουμε εμπόδια σε αυτό το brain drain που ε, παρατηρείται σε κάποιες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι αφορά τα, τα προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας και τα ε, σχετικά ταμεία. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια ε, καινοτομία στον, ε, στην σύνδεση των ταμείων έρευνας με τα ταμεία περιφερειακής συνεργασίας και συνοχής. Αυτή η καινοτομία έχουμε την ε, πεποίθηση ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και στο να κατευθύνουμε σωστά την αξιοποίηση κοντιλιών από τα διαρθρωτικά ταμεία, από τα ταμεία συνοχής, αλλά και στην εξειδίκευση της έρευνας ε, σε τομείς που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ένα τελευταίο σχόλιο για την Τρόικα και την ε, χρησιμότητά της. Ε, αντιλαμβάνεστε κύριε ότι ε, είμαστε ένα σχετικά νέο κράτος ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρό κράτος μέλος. Η ευκαιρία που είχαμε να συμμετέχουμε στο τρίο με την Πολωνία, ιδιαίτερα με την Δανία, ήταν βοηθητική στην, ε, ε, στη διαδικασία της προετοιμασίας μας για ανάληψη της ε, Προεδρίας, τουλάχιστον στο αρχικό ε, στάδιο. Ε, στην πορεία έχω την εντύπωση ότι είναι η συνεργασία με όλους τους θεσμούς και όλες τις συνιστώσεις που πραγματικά βοήθησε την, μας βοήθησε να αντεπεξέλθουμε στους ε, στόχους της ε, Προεδρίας παρά το τρίο από μόνο του. Ε, ο θεσμός, όπως ξέρετε, έχει πολλές αδυναμίες, έχει και πλεονεκτήματα. Κάθε φορά που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αλλαγή θεσμών, έτσι έχουμε την τάση να περιπλέκουμε τα πράγματα παρά να τα απλοποιούμε. Ε, δεν είμαι βέβαιη πώς θα μπορούσαμε να χειριστούμε αυτή τη σχέση μεταξύ της εναλλασσόμενης προεδρίας ε, καλύτερα. Είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε, είμαι βέβαιη, πολλές φορές και στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, ξέρω ότι είναι ε, οι τελευταίες ώρες ε, πριν να ε, πάρει ο καθένας το δρόμο του για να κάνει γιορτές με την οικογένειά του και ευχαριστώ γιατί είσαστε εδώ ε, και να ευχηθώ έτσι μια πολύ δημιουργική παραγωγική συνεργασία με, στους επόμενους μήνες ε, του Κοινοβουλίου με την Ιρλανδική Προεδρία για τους ε, σκοπούς που όλοι μαζί έχουμε θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία, Υπουργέ, ο κύριος Οντί θέλει να κάνει μια τελευταία παρατήρηση. Λοιπόν, στη Γαλλία ποτέ δεν παίρνει το λόγο κανείς μετά την, ε, τον, τον Υπουργό, αλλά τέλος πάντων επιτρέψτε μου μία παρατήρηση ότι μιλήσατε ότι είσαστε μία μικρή χώρα. Ποτέ στην Ευρώπη δεν έχουμε μικρές και μεγάλες χώρες. είμαστε όλοι καλοί Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ την Υπουργό για την παρουσία, η παρουσία της. Ευχαριστούμε για την ε, ε, παρουσίαση που έκανε, τόσο λεπτομερή. Ευχαριστώ